στο Σιάν Σαντιρέκ μπορεί να βρείτε το κείμενο αυτό. Αυτό για τα διορθωτικά. Και τώρα. Έχω και άλλες ανακοινώσεις κυρίε και κύριοι. Στις 22 Νάτου έγινε κάτι πάρα πολύ σημαντικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την 66η Γενική Συνέντευξη του ΟΗΕ, διότι για πρώτη φορά για πρώτη φορά λέγω ο μόνος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μίλησε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις 21 του. εκτελέστηκε ο Τρόι Ντέιβις. Θεωρούμε ότι η θανατική ποινή είναι κάτι το απάνθρωπο και απαράδεκτο. Και από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εμεί δηλώνουμε αντίθετη στην θανατική ποινή. Έχουν πάρα πολλέ φορέ τοποθετηθεί κατά της θανατικής ποινής ανεξαρτήτως ε, ε, ποινών που επιβάλλονται σε χώρες δημοκρατικές ή σε χώρες σαν το Ιράν όπου την ίδια ημέρα ένας 17χρονος Αλή Ρεζά Σουλτάν ε, ε, διαπαγωνισμού. Οπότε ε, θεωρούμε ότι πρόκειται εδώ περί κατάφορας παρέμβασης του, του, διεθνούς δικαίου μια που εξετελέστε ένας ανήλικος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παγίως είναι κατά της θανατικής ποινής ήταν και θα είναι. Θεωρούμε ότι έτσι δεν απονέμεται δικαιοσύνη. Τέλος, έχουμε άλλη μια ανακοίνωση η οποία αφορά την τρέχουσα στην του Κοινοβουλίου που θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική. Αυτή η εβδομάδα είναι κρίσιμη διότι πρόκειται να ψηφίσουμε την ε, δέσμη μέτρων ε, που αποτελούν ένα μεγάλο θρίαμβο, μια μεγάλη νίκη για μας. Διότι πετύχαμε να καταδείξουμε ότι η κοινοτική μέθοδος είναι η πιο δόκιμη μέθοδος ώστε κανείς να μπορεί να αντιμετωπίσει την κρίση. Όμως είχαμε κάποιες επιτυχίες διαπραγματεύσεις επίσης, οι οποίες διήρκεσαν ένα χρόνο. która powinna skrócić dotychczasową οπότε αυτή την εξαπλίδεση μέτρων θα πρέπει να την γιορτάσουμε, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι θα πρέπει να βρεθεί μια ταχυτέρα διαδικασία που να διεκπεριώνει καλύτερα σε τέτοιου είδου περιστάσει. Θα πρέπει οι νομοθέτε να ενεργούν ταχύτερα. Βεβαίω, αυτό το οποίο θέλω να πω δεν, δεν καταδικάζει ε, όλε μα τι πράξει. Απλώ σε ορισμένε περιπτώσει ισχύει αυτό. Οπότε, αυτό το οποίο θέλω να γίνει είναι να διεξαγάγουμε κάποια συζήτηση σε επαφή με του πρόεδρου των ε, πολιτικών ομάδων και να το συζητήσουμε αυτό. Και επίση να δούμε τι θα γίνει και με τους πρόεδρους των, ε, των μονίμων ε, κοινοβουλευτικών μας επιτροπών, ε, εκεί που υπάρχει πιο πολύ νομοθετική δουλειά, και να δούμε αν μπορούμε να βρούμε μια σχετική διαδικασία. Αλλά το λέω σε αυτή τη φάση απλά ως μια πρόταση. Επίσης σας υπενθυμίζω ότι την Τετάρτη ο πρόεδρος Μπάρζο πρόκειται να έρθει και να παρουσιάσει τα της κατάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μας μιλήσει και θα παρουσιάσει το πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και επίσης θα πρέπει να προσδοκούμε περαιτέρω νομοθετικές προτάσεις όσον αφορούν την αντιμετώπιση της κρίσης. Θα πρέπει επίσης να προβούμε σε ταχεία θέσπιση νομοθεσία του, ώστε να μπορέσουμε να ανασχέσουμε αυτή την πολιτική κρίση και να μπορέσουμε να, να, αντιμετωπίσουμε και την κατάσταση στην αγορά. Επίση, θα πρέπει να σταθεί ένα μήνυμα στου λαού τη Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η κοινωτική μέθοδο είναι αποτελεσματική και ταχεία στον αντιμετώπιση των καταστάσεων. Οπότε θα πρέπει να σα υπενθυμίσω ότι αύριο για πρώτη φορά θα ε, έχουμε εδώ τον Ζων Κλοντ Γιούγκερ, τον πρόεδρο του Eurogroup και θα συζητήσουμε ότι υποβάλλουμε ερωτήσει. ε, μέχρι σήμερα. Έχουμε διεξαγάγει αυτή τη διαδικασία προ τον πρόεδρο τη Επιτροπή, την αντιπρόεδρο Άστον, οπότε αυτό είναι ένα νέοτερισμό. Ε, Πρόκειται για μία νέα διαδικασία, ούτως ώστε να μπορούμε να εκπροσωπήσουμε τους συμπολίτες μας ε, σε αυτήν την αντιμετώπιση της κρίσης. Θα έρθει βέβαια και η Αντιπρόεδρος ε, Άστονη ε, στην αυριανή συζήτηση και θα λάβει μέρος και θα συζητήσουμε τα, τις ε, ε, σχέσεις, εταιρικές σχέσεις όσον αφορά την συνάντηση κορυφής της Βαρσοβίας. Οπότε, συνάδελφοι, παρακαλώ να συμμετάσχετε εις αυτές τις συζητήσεις. Πρόκειται για συζητήσεις πάρα πολύ σημαντικές από πάσης πλευράς και θα θέλαμε επίσης να ε, γίνει μια συζήτηση σοβαρή μια που αυτά είναι τους συμπολίτε μας και θα πρέπει να δείξουμε σε αυτούς ότι ενδιαφερόμαστε και ότι είμαστε δυναμικοί σε αυτές τις συζητήσεις. Αυτό σας παρακαλώ να το πράξετε, σας παρακαλώ